Επαναλαμβάνονται συνεδρίαση και τα πρακτικά της θεσινής συνεδρίας έχουν διανεμηθεί. Αν δεν υπάρξουν παρατηρήσεις, θεωρείται πως τα πρακτικά εγκρίνονται. Σύμφωνα με την ημερήσια